Τη Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωση ελέγχου βάση επιδόσεων στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική. Τέσσερα λεπτά συγγητή μα. Αξιότιμο πρόεδρε, αντιπρόεδρε, τίμα μας. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότητα 40 εκατομμύρια συναλλαγές ε, ελέγχοντάς και άλλες συναλλαγές στην ΚΑΠ κοστίζει 4 δις ετήσια καθώς οι κανόνες και οι διατάξεις που αφορούν την ΚΑΠ έχουν γίνει ακόμα πιο περίπλοκες, σύνθετες ε, και πολύπλοκες, αναμένεται ότι το κόστος ε, της εποπτείας θα είναι 58 δις σε σχέση με τον προϋπολογισμό και θα αυξάνεται το κόστος αυτό αν δεν γίνει τίποτα. Εκτιμούμε ότι 4 δις λοιπόν είναι το εκτιμόμενο κόστος ε, στο επίπεδο κράτους μέλους. Βλέπουμε ότι είναι ατέλειωτη, ατέλειωτο χαρτοβασίλειο και η γραφειοκρατία και έχουμε όλο και πιο περίπλοκες διατάξεις και σύνθετες διατάξεις ε, ένας ε, Φινλανδός γεωργός ε, κατέδειξε το παράλογο του θέματος ε, αναφερόμενος στις επίσημες αιτήσει και τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται από τις εθνικές αρχές. 33 μέτρα μήκος είχαν τα έγγραφα αυτά. Είναι περίπου το μήκος δύο πλήρων γραμμών ε, των θέσεων των Ευρωβουλευτών στην Ολομέλεια και αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και δεν ε, γίνουμε πιο αποτελεσματικοί ανακουφίζοντας ε, το βάρος ε, των αγροτών, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει νέο αίμα το οποίο θα εισαχθεί στη γεωργία με νέους γεωργούς. Δεν είναι όμως μόνο θέμα της γεωργίας αυτό. Περίπλοκοι κανόνες και διατάξεις σημαίνουν αναπόφευκτα ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν δαπανώνται αποτελεσματικά. Ακόμα χειρότερο από την αναποτελεσματικότητα είναι η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για τη σωστή χρήση των κονδυλίων βλέπουμε ότι ίσως σε κρατική ελέγχη θα μπορούσαν να προσφέρουν μια λύση. Η έκθεση λέει ότι σε σχέση με τις επιδόσεις και τους ελέγχους θα πρέπει η ποιότητα κυρίως να αναβαθμιστεί όσον αφορά τους ελέγχους στο επίπεδο των κρατών μελών. Αποτελεσματικότητα, συνεκτικότητα και συνάφεια και σωστές αλλαγές. Για να ανακουφιστεί το βάρος για τους εποφελούμενους οι αρχές θα πρέπει να διοργανώσουν επιτόπου ελέγχους με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνονται οι γεωργοί με πολλαπλούς ετήσιους τέτοιους ελέγχους από τις Εθνικές Αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελεγκτικό συνέδριο. Θα πρέπει λοιπόν η ενιαία λογιστική ε, διαδικασία να εφαρμόζεται όσον αφορά τους ελέγχους. Θα πρέπει επίσης σε σχέση με τον, ε, την ταυτοποίηση των καλύτερων επιδόσεων και των χειρότερων επιδόσεων όσον αφορά κράτη-μέλη, εκείνα που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις πρέπει να μπορέσουν να, ε, να αντιμετωπίζουν λιγότερους τέτοιους ελέγχους από ότι οι χειρότεροι. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα αυτής της προσέγγισης είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ώστε να μπορούν οι, ε, τα κράτη που έχουν τις χειρότερες επιδόσεις να υποφεληθούν. Απλούστευση λοιπόν είναι κάτι το αναπόφευκτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε αυτή την πορεία και θα πρέπει να συνεχιστεί η πορεία αυτή. Από πλευράς εισηγητού στόχος είναι να μπορέσουν να ανακουφιστούν οι γεωργοί και ταυτόχρονα να παράσχουμε καλύτερους ελέγχους όσον αφορά τα χρήματα των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye, το οποίο θα κρατήσει πέντε λεπτά. Για ένα, λεπτά, για ένα λεπτό, ο κυρία Ναβακόβα, παρακαλώ. Ο κύριος Ναβακόβα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η καλύτερη πολιτική δημοσίων σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν ακριβώς να προβάλλουμε περισσότερο τις ε, επιδόσεις, τα αποτελέσματα θετικά που πετύχαμε από κοινού Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι ο κύριος Πέτρης Σαρβαμά έχει ε, συντάξει μια εξαιρετική έκθεση και νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από την έκθεσή του αυτή. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές η έλεγχη γεωργική είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική, ιδιαίτερα επαχθής για τους γεωργούς. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιταχύνουμε όλες τις σχετικές διαδικασίες. Όσον αφορά δηλαδή τις πληρωμές και όσον αφορά όλες τις άλλες πτυχές διαδικασίας. Και οι γεωργοί οι οποίοι έχουν καλές επιδόσεις θα πρέπει να ελέγχονται όλο και λιγότερο και βέβαια να ισχύει και το αντίστροφο. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα επιβράβευσης και προφανώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες ψηφιακές τεχνολογίες. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουμε την εργασία μας και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις συγκεκριμένων γεωργικών εργασιών. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια των δύο μεταρρυθμίσεων της κοινή γεωργικής πολιτικής είδαμε τελικά ότι τα μέτρα γίνανε πιο πολύπλοκα και τερογενή. Και βλέπουμε ότι βαρύνουν αυτή τη στιγμή τους γεωργούς και έχουμε και περισσότερα σφάλματα. Προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής χρειάζεται μία απλούστευση και μείωση της γραφειοκρατίας. Να μειωθεί το κόστος των ελέγχων που όπως μας είπε ο συγητής είναι ήδη 4 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης οι υπηρεσίες πληρωμών θα πρέπει να λειτουργούν με έναν νέο τρόπο προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος, το οποίο έχει εντοπίσει σε 42 συγκεκριμένου οργανισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά για να σας παρακολουθούν και διερμηνείς. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε πολιτικές προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις στις εσφαλμένες δηλώσεις που κάνουν ορισμένες υπηρεσίες πληρωμών. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν κοινά κριτήρια για να δούμε ποια κράτη-μέλη έχουν τις καλύτερες επιδόσεις και ποια είναι τα κράτη-μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο τις βέλτιστες πρακτικές. Με άλλα λόγια χρειαζόμαστε μια εξορθολογισμένη νέα κοινή γεωργική πολιτική που θα στρέφεται όλο και περισσότερο προς τους αγρότες και τους γεωργούς. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πετύχουμε του στόχου μα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω την πρωτοβουλία αυτή και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα απλούστευσης της ΚΑΠ είναι σημαντικό να είναι αυτό επωφελές ε, όχι μόνο για τους γεωργούς αλλά και εκείνους ε, που η επιβίωσή τους, ε, το εισόδημά τους εξαρτάται από τη γεωργία και το πρασίνισμα της γεωργίας συνδέεται με την υπεύθυνη χρησιμοποιείται από εκείνους που γενναίες επιγενεών εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι στη νέα περίοδο πολλοί κανόνες έχουν εντωμεταξύ τροποποιηθεί και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες να δραχθούν τις ευκαιρίες και να αρχίσουν με ήπια μέτρα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα της κοινή γεωργικής πολιτικής που πλήττει τους αγρότες είναι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξει απλούστευση του συστήματος προκειμένου να βελτιωθεί και να αυξηθεί η αποδοτικότητα κατά την παροχή ενισχύσεων της κοινή γεωργικής πολιτικής. παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δοθεί λύση στα μεγάλα προβλήματα της γεωργίας. στη χώρα μου την ελλάδα οι φτωχοποιημένοι από το μνημόνιο έλληνες αγρότες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά καθώς τη χρονιά που πέρασε δοκιμάστηκαν από τις καταστροφές στην παραγωγή τους που έπληξαν την πατρίδα μου ενώ η φόρο επιδρομή που βιώνουν και βίωσαν με εντολή της τρόικας επεκτάθηκε παράνομα και στις κοινοτικές ενισχύσεις που λαμβάνουν. έτσι την τελευταία πενταετία το εισόδημα των ελλήνων αγροτών μειώθηκε κατά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και οι φόροι αυξήθηκαν κατά. 150 παράλληλα η κρίση που ξέσπασε στη γεωργία λόγω του ρωσικού εμπάργου κατέστρεψε οικονομικά τους έλληνες αγρότες. για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να υπάρξει άμεση αύξηση των ενισχύσεων στους στοχοποιημένους από τα μνημόνια έλληνες αγρότες. ευχαριστώ. ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. συζητάμε ένα σημαντικότατο θέμα αλλά έχουμε ενώπιόν μας μια εξαιρετική έκθεση που συντάχθηκε από έναν εξαιρετικό συνάδελφο που άγγιξε το πρόβλημά του στην καρδιά του. χαρακτηριστικά μέσα από αυτά που είπε δεν χρειάζονται και πολλά εμείς να συνεισφέρουμε και να προσθέσουμε. Αναφέρομαι στη λέξη αποτελεσματικότητα. Και αυτή αποδίδεται όταν έχεις ενώπιό σου το κάδρο του προβλήματος, που είναι 50 εκατομμύρια πράξεις, που είναι έλεγχοι που κοστίζουν 4 δισεκατομμύρια, που ουσιαστικά αντιστοιχούν στο 7% των χρημάτων που δίνουμε για την κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή κάθε 100 ευρώ που δίνουμε, τα 7 πάνε αποκλειστικά και μόνο για ελέγχους και αν πραγματικά δεν είμαστε διατεθειμένοι να αξιοποιήσουμε αυτή τη σημαντική έκθεση και να λύσουμε στη ρίζα του το πρόβλημα και η αγροτική οικονομία θα πλήττεται οι αγρότε μα θα ταλαιπωρούνται και κερδισμένοι θα βγαίνει και πάλι η γραφειοκρατία η οποία σκοτώνει κάθε προοπτική και κάθε ανάπτυξη. Είναι ευκαιρία λοιπόν να στηρίξουμε του αγρότε μα καταργώντα τον διοικητικό φόρτο και δίνοντα και θα εισηγηθώ μια καινοτόμα πρόταση δίνοντα τη δυνατότητα αυτοελέγχου σε αυτά τα οποία γίνονται στο γεωργικό τομέα. Η απλούστευση είναι ένας τρόπο για να περιορίσουμε τον αριθμό των επιτοπίων ελέγχων απλούστεροι κανόνες. Ε, τι σημαίνει αυτό, ότι θα είναι ευκολότερη η εφαρμογή τους, ευκολότερο να δουλεύουν με βάση αυτών των κανόνων οι γεωργοί και ευκολότερη και η έλεγχη από, για τις αρχές. Όπως είπατε, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με την άσκηση απλούστευσης όπως είπατε, και έχουμε λάβει ε, τα σχόλια πολλών εμπλεκομένων φορέων. Έχουμε ήδη εφαρμόσει κάποιες αλλαγές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει και άλλες προτάσεις στους επόμενους μήνες. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε νέου κανόνε όμω για να επηρεάσουμε τον αριθμό των ελέγχων με του οποίου πρέπει να αντιπεξέλθουν οι γεωργοί βάσει των ε, κανονισμών. Μπορούν τα κράτη-μέλη με αξιόπιστα συστήματα διαχείριση και ελέγχου να περιορίσουν τον αριθμό των επιτοπίων ελέγχων και κάποια κράτη-μέλη έχουν ήδη εκφράσει την ενδιαφέρον του να χρησιμοποιήσουν αυτή τη ε, δυνατότητα που του δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεργαζόμαστε στενά μαζί του ε, ούτω ώστε να πληρούνται όλε οι προποθέσει για αυτή την ευκαιρία καλύτεροι κανόνες, καλύτερη εφαρμογή, καλύτερη επίσης εκλασιμότητα, τόσο ώστε να ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει κατασπατάληση του δημοσίου χρήματο. Ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη βάσει τη κείμενη νομοθεσία να οργανώνουν του ελέγχου με τρόπο ώστε να περιορίσετε το άχθο για του γεωργού. Να μην ξεχνούμε όμω ότι μόνο 5% των γεωργών ελέγχονται επιτόπου για την συμμόρφωση με του ελέγχου κοινή γεωργική πολιτική. Ε, Ω επιτοπλίστων, ε, οι ελέγχοι απορρέουν από εθνική νομοθεσία και από του κανόνε τη πολλαπλή Αυτό όμω δεν προκύπτει από την νομοθεσία που σχετίζεται με την κοινή γεωργική πολιτική, για του γεωργού. Φυσικά δεν έχει καμία σημασία ή το έλεγχο έρχεται από, το, την από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το ε, κράτο μέλο. Ε, θέλουν λιγότερου ελέγχου και δίκιο έχουν. Δεν πρέπει να ασχολούνται με την γραφειοκρατία, αλλά με το να καλλιεργούν τα χωράφια του. Και πιστεύουμε τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα για να ομαδοποιήσουν του ε, δικού του ελέγχου με αυτού που ε, προκύπτουν από τι υποχρεώσει που έχουν αναλάβει στα πλαίσια τη κοινή γεωργική και θα ήταν γι' αυτό καλύτερο να γίνεται αποτελεσματικότερη ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Φυσικά παραμένουν απαραίτητοι οι έλεγχοι αν έχουμε ε, επιπρόσθετες ε, ε, προϋποθέσεις για να χορηγηθεί μια επιδότηση, τότε συνεπάγεται αυτό και ελέγχους και όσο περισσότερες είναι οι απαιτήσει, τόσο περισσότεροι και περίπλοκοι είναι οι έλεγχοι. Φυσικά όλοι έχουν το δικαίωμα να ξέρουν αν υπάρχει σωστή χρήση των κονδυλίων μέσω των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα απορρίψουμε οποιαδήποτε πρόταση αντιβαίνει ε, στην λογική της ε, χρήστης ε, διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν το ποσοστό λάθος το 2% είναι το κατάλληλο σημείο σύγκρισης για μια τόσο περίπλοκη πολιτική όπως η κοινή γεωργική πολιτική και συγκεκριμένα για την πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο κόστος και το όφελος ε, των ελέγχων θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και αυτή τη διάσταση, αλλιώς ε, θα χάσουμε την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε αποτελεσματικά την κοινή πολιτική. Είναι ο κρογωνιαίος λίθος, ήταν και παραμένει ο κρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκή Ένωσης η κοινή πολιτική και είναι καθήκον μας να μεριμνήσουμε ώστε να είναι αποτελεσματική αυτή η πολιτική και να συνιστά ε, σημείο στήριξη ε, για τους πολίτες αλλά και για τους γεωργούς. Οι φορολογούμενοι θέλουν να είναι σίγουροι ότι υπάρχει μια χρηστή διαχείριση των των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα ευχαριστώ τον κύριο Σάβαμαρ ε, για την έκθεσή του. Ε, είναι άλλη μια συμβολή στην πρώτη συζήτηση για την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Κλείνει η συζήτηση και αύριο θα ψηφίσουμε. Τώρα, συνάδελφοι,